Good afternoon, ladies and gentlemen. σας απόγευμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και ευχαριστώ ιδιαίτερο στις και τους συναδέλφους που έχουν προσέλθει σήμερα. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Θα περιμένουμε να εμφανιστούν αργότερα οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας στη διάρκεια των συζητήσεων. Η συνεδρίασή μα είναι αφιερωμένη σε δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες για άλλε επιτροπές, για γνωμοδοτήσει μάλλον. Το ένα για την νομοθεσία για το ΠΔΠ. Η πρώτη γνωμοδότηση πηγαίνει στην Επιτροπή Μεταφορών και αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, δηλαδή τα λεγομενα ten t ten 10TAF. Το δικό μας ενδιαφέρον έγκυται στην σημασία των δικτυων ten 10TAF για την βιώσιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την σύνδεση μεταξύ πολιτικής συνοχής και πολιτικής μεταφορών όταν συζητήσαμε την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και τους οριζόντιους κανονισμούς. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Ο προτινόμενος κανονισμός συμβάλλει στην εκπλήρωση του βασικού στόχου να γίνουν οι μεταφορές ασφαλέστερες, πιο προσβάσιμες και καθαρότερες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας. Ο γενικός στόχος της πρότασης της Κομισιόν είναι να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις και το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας που επηρεάζει την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Επομένως υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που εστιάζει η πρόταση, όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση του συντονισμού κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για διασυνοριακά έργα, ο καθορισμός προθεσμιών στους κανόνες για τη χορήγηση αδειών και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θέλουμε να τονίσουμε ότι το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών έχει ζωτική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης και συνολικά ωφέλει στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω των αρχικών τροπολογιών που κατέθεσα στην πρόταση εκ μέρους της Επιτροπής ΡΕΤΖΙ, ήθελα να δώσω έμφαση στα εξή σημεία. Πρώτον, διασφάλιση των περιβαλλοντικών πτυχών κατά το σχεδιασμό και εφαρμογή του TNT. Συγκεκριμένα, προώθηση μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και επίτευξη στόχων χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, εκτός από τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, απαιτείται εντελεχής αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων όσον αφορά την απασχόληση, την υγεία, μείωση των ατυχημάτων, την ποιότητα ζωής, τα τοπικά ωφέλη και την κοινωνική ένταξη. Δεύτερον, αναφορά, σαφής αναφορά ότι το TNT θα λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις γειτονικέ παραμεθόριες περιοχές, συμβάλλοντας περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα αυτών των περιοχών. Τρίτον, διασφάλιση της αποτελεσματικής συμβολής των έργων του TNT στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Σε αυτό θα συμβάλλει κατά ένα μεγάλο βαθμό κοινωνικός διάλογος και ο διάλογος με τους πολίτες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αυξάνοντας την αίσθηση του κοινού καλού για τα έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών και της αξιοπιστίας. Τέταρτον, θέτω επίσης το θέμα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών θα χαρώ να λάβω και από τους συναδέλφους τις προτάσεις τους για τροπολογίες. Να σημειώσω επίσης ότι για διαδικαστικού λόγους η τροπολογία 5 έχει αποσυρθεί. Θα καταθέσω νέα τροπολογία στο ίδιο πνεύμα, εκφράζοντας αντίθεση στη μείωση του προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής μέσω της συνεισφοράς του ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τιμές 2018 στη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Thank ευχαριστώ κυρία Παπαδάκη. Ο σκιώδης εισηγητής κύριος Βαλκάρσελ Σίσο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιθυμώ να ευχαριστήσω για τις τροπολογίες. Αξίζει τον κόπο να γίνει προσπάθεια βελτιώσεως του κειμένου. Θα ήταν δυνατόν να προσθεθούν και άλλες τροπολογίες έτσι ώστε να ενισχυθεί η βασική αντίληψη, το κόνσεπτ δηλαδή, ότι οι συνδέσεις δεν πρέπει να εξυπηρετούν μόνο τις ε, ορεινές περιοχές, αλλά όλες τις ε, μειονεκτικές περιοχές, όλες τις μειονεκτικές περιφέρειες και να τονίζουν συνέργειες για την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς παρακαλώ. Κύριε Ζέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ εγκαρδίως και τον εισηγητή για την σύνταξη της πολύ σημαντικής αυτής γνωμοδότησης. Πώς θα ενωθεί η Ευρώπη χωρίς δίκτυα μεταφορών και να σκεφτούμε ιδίω το σιδηροδρομικό δίκτυο και ιδίω των υψηλών ταχυτήτων διότι μιλούμε συχνά και πολύ για προσπάθεια μείωση των διοξιδίων του άνθρακο και μείωση άλλων επιβλαβών εκπομπών αερίων. Εκεί μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αν δούμε όμω την εξέλιξη στην Ευρώπη θα δούμε ότι συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή αυξάνονται όλο και περισσότερο οι μεταφορές με φορτηγά αυτοκίνητα, όλο και περισσότερο οι εναέριε μεταφορές, απόλυτη στασιμότητα για να μην πω και υποχώρηση στον σιδηρόδρομο. Και μία από τι συνέπειε είναι επίση, μάλλον ένα από του λόγου, είναι ότι παρόλες τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές σχεδιάσεις για τη δημιουργία ενός σιδηροδρομικού δικτύου δεν έχει και καταστεί δυνατόν να υλοποιηθεί. 23,7 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν προβλεφθεί για τα τρένα μεγάλης ταχύτητας και έγιναν και κάποια πράγματα αλλά και αυτό σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε από το ελεγκτικό συνέδριο πολύ πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, οι χώρες μέλη ανέπτυξαν σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας, αλλά μόνο εσωτερικά μέσα στις ίδιες τους τις χώρες. Όπου επρόκειτο για διάβαση μεθορίου δεν έγινε σχεδόν τίποτα ή πάντως πάρα πολύ λίγα πράγματα. Πολύ συχνά σταματούν 15-20 χιλιόμετρα από τα σύνορα για την επόμενη χώρα, τη γειτονική τους χώρα. Και δεν επιτρέπουν να γίνει έργο που να διαβαίνει τα σύνορα. Θεωρώ ότι πρόκειται για απολύτως απαράδεκτη κατάσταση. Και μια προσπάθεια που γίνεται με εναρμόνιση των προτύπων και προδιαγραφών μέσω του πακέτου σιδηροδρόμων για να υπάρξει επιτέλους και στην Ευρώπη ένα ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο και τέτοιες προσπάθειες λοιπόν εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο των συζητήσεων που διαρκεί εδώ και χρόνια. Κάθε χώρα μέλος προσπαθεί να παίξει με τα τρενάκια της μέσα στην επικράτειά της με κάποια μέτρη επιτυχία. Αλλά παρόλη την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που υποτίθεται ότι θα επιτευθεί δεν έχει γίνει. Δεν έχουμε καταφέρει να ξεφύγουμε από κάποια πρώτα διστακτικά βήματα. Άλλε χώρες, μεγάλε δυνάμεις όπως η Κίνα προσπαθούν τώρα μέσα στα πλαίσια αυτού του One Road, One Belt να προχωρήσουν. Έχουν πάει, έχουν πιάσει λιμάνια και της Ευρώπης και προσπαθούν τώρα προωθώντα επενδύσεις και στον σιδηρόδρομο να προωθηθούν να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ενώ ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός ακόμα υστερεί. Ζητήσω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα την προτρέψω να ενισχύσει τις προσπάθειες και να σκληρύνει τη στάση της εκεί όπου οι χώρες μέλη δεν τηρούν τους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς και δεν προωθούν κοινό ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο να τους δείξει την βούλησή της ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να ξεπεραστούν τα σημεία εχμής όπου δεν συμβεί αυτό να τους κόψει τις επιδοτήσεις. Διότι χρειάζεται επιτέλους να υπάρξει έντιμη συνεργασία για να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά που εμποδίζουν το διαμεθοριακό εμπόριο. Έχουμε την ευκαιρία και τώρα, όταν θα συζητήσουμε τους νέους κανονισμούς, να καταστήσουμε το μήνυμα αυτό σαφές. Και νομίζω ότι η έκθεση του Έλληνα, λέει, συναδέλφου μας, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο τώρα στον, στην εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Βερσίνη, DG Home. Δεν είναι παρόν όμως, διότι όλοι έχουν πάει τώρα στην Επιτροπή Περιφερειών στην <clears throat> Ευρωπαϊκή, δηλαδή Επιτροπή Περιφερειών και δεν είναι εδώ, στην Περιφερειακή δική μας Επιτροπή. Καλώς, δεν έχουμε άλλον που να ζητεί να συμμετάσχει στη συζήτηση. Θα προτείνουμε λοιπόν, θα προτείνω μάλλον, προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών την 3η 16 Οκτωβρίου, 16 Δεκάτου, το μεσημέρι, για τροπολογίες, ξαναλέω. Αυτό θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Ρέτζι στις 15 Ενδεκάτου Νοεμβρίου. Και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Τραν προβλέπεται στις 3 Δωδεκάτου Δεκεμβρίου. Άρα θα είμαστε απολύτως μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Τώρα, το επόμενο. Α, με συγχωρείτε ένα λεπτό, με συγχωρείτε ένα λεπτό, λέει Αυτά σχετικά με τη γνωμοδότηση του κ. Παπαδάκη. Τώρα, η επόμενη γνωμοδότηση θα παρουσιαστεί από τον συντάκτη της κ. Μίλτενμπουργκ, ο οποίος έρχεται, είναι καθοδόν από μία αίθουσα σε άλλη. Βλέπω ότι και ο κύριος Γκάμπελικ είναι, η κυρία μάλλον Γκάμπελικ είναι παρούσα, σκιώδη συγγήτρια. Μπορούμε να αρχίσουμε την ε, συζήτηση. Έχουμε εκπρόσωπο της ε, Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμών της Επιτροπής. Α, ωραία, χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ό,τι συνήθω σήμερα. Ναι. Βεβαίω, να περιμένουμε λίγα λεπτά. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Σας ευχαριστώ. Θα περιμένουμε την έλευση του κυρίου Ματέη Βαν Μίλτενμπουργκ.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 Χαίρομαι που σας βλέπω κύριε Μίλτενμπορκ. Βεβαίως όλοι κινούμεθα από μια συνεδρίαση σε άλλη. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. περιμέναμε λίγο για να έλθετε, για να μπορέσετε να παρουσιάσετε την γνωμοδότησή σας για το κράτος δικαίου, για θέματα δηλαδή κράτους δικαίου. Έχουμε τη σκιώδη συγκήτρια, έχουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε αμέσως, κύριε Βαν Μίλτεμπορντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας. Γιατί πραγματικά είναι φορτωμένο το πρόγραμμα αυτές τις ημέρες και ω εισηγητή έπρεπε να είμαι στην Επιτροπή Μεταφορών για ένα άλλο ζήτημα. Θα ήθελα όμως ε, αρχικά να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση η οποία είναι πολύ θετική κατά τη γνώμη μου. Έχει ως στόχο την προστασία του ενωσιακού προπολογισμού. Για να το πω και λίγο ομά, δεν έχει να κάνει με την επιβολή κυρώσεων στα κράτη-μέλη που δεν τηρούν το κράτος δικαίου. Πρωταρχικό στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι ε, προστατεύουμε τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, γιατί και σε αυτή την Επιτροπή, αλλά και σε άλλε, καθώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, πάντα μιλάμε για τον προπολογισμό για τα επόμενα έτη. Πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε για αυτό τον προπολογισμό και να διασφαλίσουμε και την ελοποίηση των στόχων του προπολογισμού. Δυστυχώ αυτό δεν ισχύει πάντα. Γνωρίζουμε για παραδείγματα όπου κάποιες φορές, ευτυχώς αυτό συμβαίνει κατά εξαίρεση βέβαια, για παράδειγμα μπορεί να ε, λάβει χρηματοδότηση ένα πρόγραμμα μετά από έναν ε, ψευδεπίγραφο διαγωνισμό προς ε, ημετέρους, αν θέλετε, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες. Και μετά βλέπουμε ότι δεν μπορεί ε, να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Όμως εμείς ε, που θέλουμε να φροντίσουμε για την πραγματική υλοποίηση αυτών των έργων, γεφυρών, δρόμων κτλ. Χρειαζόμαστε ομολόγους και χρειαζόμαστε και ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και όταν έχουμε να κάνουμε με τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια ευρώ, πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και τέτοιου είδου προβλήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έχουμε λοιπόν διορθωτικά τέτοια ζητήματα, προβλήματα με το κράτο δικαίου, την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, μια διορθωτική υπονόμευση τη καταπολέμηση τη διαφθορά ε, και της απάτης. Ως λύση λοιπόν ε, ε, έσχα τη ανάγκης, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να επέμβει. Επομένως, δεν έχει να κάνει όλο αυτό με την επιβολή κυρώσεων. δεν έχει να κάνει με τον μεμονωμένο φοιτητή που θέλει να πάει Εράσμου και δεν θα πάρει την υποτροφία του ή για μια μικρομεσαία επιχείρηση ε, που δεν μπορεί να λάβει μια επιδότηση έχει να κάνει με τις γενικευμένες ελλείψεις ε, στο κράτος δικαίου που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς επειδή πρόκειται για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα πίσω από τις τροπολογίες είναι ζήτημα του Συμβουλίου ε, έχουμε να κάνουμε πλέον με την εκτέλεση του προπολογισμού. Από αυτή την άποψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το πολύ συγκεκριμένο καθήκον να διασφαλίσει ε, τη σωστή ε, διαχείριση ε, και εκτέλεση του προπολογισμού. Γι' αυτό διορθώνω. Πρέπει να βγάλουμε το Συμβούλιο από τη μέση, εκτός κι αν δεχτούμε ότι παρεμβαίνει το Συμβούλιο στην εκτέλεση του προπολογισμού, αλλά τότε δεν, γίνονται σεβαστές συνθήκες. Έχουμε και το άρθρο 7 ε, και δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή άγουσα στην προηγούμενη περίπτωση. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε και να διευκρινίσουμε και προς το Συμβούλιο ότι δεν τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι το ultimum remedium που λέμε και στα λατινικά. Η λύση ανάγκες λοιπόν, όταν ε, πρέπει πραγματικά να μεριμνήσουμε για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τέλος. Όταν εξετάσαμε την έκθεση Westphal, είπαμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε την οικονομική, κοινωνική και εδαφική ε, συνοχή και σύγκληση μόνο αν τα φροντίσουμε όλα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένω, σα καλώ να καταθέσετε τροπολογίε αν το θεωρείτε απαραίτητο, αλλά να έχετε κατά νου ότι δεν πρόκειται για κάποιε τιμωρητικέ κυρώσει προ ε, κράτη-μέλη. Είναι ένα κανονισμό που θα ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη και, αν, και όποιο μάλλον σέβεται του κανόνε και το κράτο δικαίου. Δεν χρειάζεται να φοβάται ότι θα περικοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο τώρα στους Κιώδης. Ο κύριος Γκέμπερικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Βον Μίλτεμπουργκ για το σχέδιο γνωμοδότησης για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Πώς δηλαδή θα φροντίσουμε ότι ο νεσιακός προπολογισμό χρησιμοποιείται ε, σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Επειδή είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, μόνο αν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη που σέβεται το κράτος δικαίου και την ασφάλεια δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη, μπορεί να, ε, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ε, και τα ευρωπαϊκά κονδύλια τη χάνουν της επαρκούς ε, προστασία. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να υπάρχει αιρεσιμότητα ε, την οποία θα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο συνάδει και με την ισχύουσα νομοθεσία, με, το, με τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι τη βασική ευθύνη πρέπει να την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει σωστά προκαθορισμένες ε, αρμοδιότητες σε περίπτωση ενεργοποίησης του μηχανισμού. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει ε, να εκφέρει γνώμη σε αυτό το πολύ λεπτό ζήτημα του κρατούς δικαίου. Θα πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα τη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε μια ε, δίκαιη, δημοκρατική και πρακτική λύση. Επίση, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι μεμονωμένοι δικαιούχοι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν θα πληγούν από αυτό το μηχανισμό. Όπω, για παράδειγμα, οι φοιτητέ Εράσμου ή οι μεμονωμένοι ερευνητέ. Δεν γίνεται αυτοί να πλήττονται και να τιμωρούνται εξαιτία ε, ελλείψεων στο ό,τι αφορά το κράτο δικαίου στη χώρα του. Από την άλλη, είναι σημαντικό να μην υπάρχουν υπερβολικά πολλέ εξαιρέσει. Γιατί έτσι δεν θα έχει πρακτικό αντίκτυπο ο μηχανισμό και δεν θα καταφέρει να πετύχει το στόχο του. Έτσι προτείνω να μην επεκταθούν περαιτέρω οι εξαιρέσεις. Τέλος, η δυνατότητα που θα έχουμε εμείς για την ε, διαφύλαξη ε, του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά την ε, δαπάνηση ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι κάτι το οποίο μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που σέβεται το κράτος δικαίου και την ασφάλεια δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Μόνο έτσι, μόνο έτσι έχουμε τα πραγματικά εχέγγυα σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που προκύπτουν από τα χρήματα των Ευρωπαίων Φορολογουμένων. Για μα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την πρόταση ω σημαντικό μέτρο διασφάλιση ότι οι γενικέ ελλείψει στον τομέα του κράτου δικαίου δεν ε, θα γίνονται πλέον ε, δεκτέ και ανεκτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Ζωάννα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που πήραν το λόγο προηγουμένως. Ως μέλος ε, της Επιτροπής αυτής, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ζήτημα. Αυτά τα κονδύλια είναι θεμελιώδους σημασία ε, για την ανάπτυξη των χωρών αυτών, ιδίω της Ανατολικής Ευρώπης, όπου αυτά τα κονδύλια πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις έννοιες που χρησιμοποιούμε. Γιατί βλέπουμε τη δικαστική εξουσία με άλλες έννοιες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κονδύλια που φτάνουν απευθείας σε Ευρωπαίους πολίτες. Μιλούμε δηλαδή για δικαιούχους που έχουν ίσα δικαιώματα σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους πολίτες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτή βέβαια είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ακόμα και ο τίτλο ε, θεωρώ ότι δεν είναι αμερόληπτο. Προστασία του ενωσιακού προπολογισμού. Νομίζω ότι είναι λίγο περιβολικό αυτό. καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να οριστεί σαφώς και επαρκώς. Υπάρχει σαφής όμως ορισμός ε, της ασφάλειας, του κράτους δικαίου μάλλον. Έχουμε συμφωνήσει όλοι για τις αρχές που θα πρέπει να τηρούνται. Είμαστε δηλαδή πολύ αυστηροί με τα κριτήρια ε, που θα επηρεάσουν άμεσα αυτό τον ορισμό. Τι είναι λοιπόν το κράτος δικαίου, ποιος το προσδιορίζει και με ποιον τρόπο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Mr. Deutsch, you have the floor. Κύριε Deutsch. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις σκέψεις μου για το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο κανονισμού για θέμα για το οποίο γίνεται πολύ έντονη πολιτική συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στον έξω κόσμο. Δεν θα πρέπει να παριστάνουμε ότι δεν το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Ξέρω ότι ο εισηγητής δεν τοποθετήθηκε πολιτικά, δεν πήρε θέση ε, όσον αφορά αυτή την πολιτική συζήτηση. Ήθελα απλώς να το επισημάνω αυτό το στοιχείο. Δεν θέλω να ε, μπω σε πολιτική συζήτηση, αλλά θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω ότι ε, πρόκειται για ένα πολύ καυτό πολιτικό ζήτημα ταυτόχρονα. Δεν συμφωνώ με τη δήλωση ότι το σχέδιο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλό σχέδιο ε, ε, κανονισμού. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει πολλές τόσο κακές προτάσεις σαν αυτή που έχουμε ε, μπροστά μας. Ε, πρέπει να σας πω ότι από νομικής απόψεως είναι κάτι το ε, απίθανο. Ένας ένα θεσμικό όργανο που υποτίθεται ότι προστατεύει το κράτος δικαίου να ενεργεί κατά των αρχών του δικαίου. Δεν είναι αυτό αυτό το νόημα της δημοκρατίας του 21ου αιώνα ε, όταν ε, μιλάμε για τις ευρωπαϊκές αξίες. Δεν είναι δυνατόν ε, να μην ορίζεται σαφώς το κράτος δικαίου ή οι ορισμοί που χρησιμοποιούμε να είναι πολύ ελαστικοί και να χρησιμοποιούνται για να αιτιολογήσουν οποιαδήποτε θέση και να δημιουργούν μια κατάσταση ε, ανυπόφοροι. για τα θεσμικά όργανα. Αν διαβάσει κανείς αυτό το σχέδιο, θα δει ότι δεν περιλαμβάνει κανονισμούς που να αξίζουν το όνομά τους. Και επίσης θα ήθελα να υποστηρίξω ότι αν η πρόταση αυτή δεν αφορά κυρώσεις, τότε κάποιος που έχει λίγη πείρα από, τις, από την περιφερειακή πολιτική, και εγώ είμαι εδώ 9 χρόνια, ε, ας μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι οι επιπλέον αρμοδιότητες που δίνει ο κανονισμός αυτός σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Δεν θα πρέπει να παριστάνουμε ότι τι, τι θέλουμε να πούμε δηλαδή, ότι δεν υπάρχει ενισχύ νομοθεσία που να επιβάλλει κυρώσεις όταν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας. Φυσικά, οι ε, Φυσικά υπάρχουν άλλες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι καθαροί συνεισφορείς και άλλοι που είναι καθαροί ε, λήπτες κονδυλίων. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά υπάρχει ένα σύστημα που εφαρμόζεται στην πράξη και υπάρχουν κανόνες για τις ε, κυρώσεις που επιβάλλονται. Όλα τα κράτη-μέλη που παίρνουν ε, κονδύλια στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής, υπάρχονται σε κάποιοι κανόνες και υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν διαδικασίες ε, Επιβολή κυρώσεων εναντίον ε, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και οποιοδήποτε άλλου. Υπάρχει ένα σύστημα που λειτουργεί, ενισχύει. Τι θέλουμε να πετύχουμε παραπάνω με αυτό το σχέδιο κανονισμού. Και όταν πρόκειται για ένα σχέδιο που δεν πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, τις νομοθετικές, ε, ένα τέτοιο σχέδιο έχουμε μπροστά μας, και ταυτόχρονα αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, αν υπάρχουν παραβάσεις ε, ε, ή οτιδήποτε τέτοιο, υπάρχουν κυρώσεις που προβλέπονται από το ισχύον σύστημα. Το άλλο μου επιχειρήμα απευθύνεται και πάλι στην Κομισιόν και όχι στους συναδέλφους εδώ. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό Γιατί ενώ η νομοθεσία λέει ότι οι τελικοί δικαιούχοι δεν θα πρέπει να υφίστανται τις επιπτώσεις ε, της κακής διαχείρισης. Αυτό είναι το νόημα της ε, επιμερισμένης διαχείρισης. Έτσι χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Αν υπάρχει ένα έβριμα που δείχνει ότι συστημικά δεν ε, ε, γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου, ακόμα και τότε δεν μπορεί να υποστεί ε, ένα μειονέκτημα λόγω αυτού ο τελικός δικαιούχος. Η Κομισιόν δεν θα μπορέσει να επιβάλλει κυρώσεις στην περίπτωση αυτή. Οπότε όλη η έννοια του share management, της επιμερισμένη διαχείρισης, χάνει τη λογική της. Γιατί από το σημείο αυτό και μετά θα είναι οι ε, γραφειοκράτες της Βρυξέλλες που θα αποφασίζουν ποιοι ε, δρόμοι στη Ρουμανία ή ποια αναπτυξιακά προγράμματα στη Γερμανία ε, αξίζει να πάρουν ενισχύσεις και γενικά πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια της περιφερειακής πολιτικής. Και δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Ε, στο χαρτί μπορεί να γράψει κανείς ό,τι θέλει, αλλά δεν θα περάσει τη δοκιμασία της πραγματικότητας. Είναι αδύνατον να παρακάμψει κανείς τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και να δώσει τα χρήματα κατευθείαν στους δικαιούχους κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει, στην, ε, υπάρχει μια ιστορία που λέμε στην Ουγγαρία ε, σχετικά με μαθητές, ένα ανέκδοτο τέλο πάντων που καταλήγει στο ότι αυτό το ζώο δεν υπάρχει. Ε, περί αυτού πρόκειται. Αυτό το ζώο για το οποίο μιλάμε εδώ δεν υπάρχει. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε αναλάβει μια ανέφικτη αποστολή. Mission impossible. Ε, σαν πολιτική βέβαια συχνά αναλαμβάνουμε τέτοιες αποστολές και δεν θέλω να αμφισβητήσω τις καλές σας προθέσεις αλλά έχω πολύ αρνητική γνώμη για αυτό το σχέδιο ε, κανονισμού. Η κυρία Κρέλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Παρακολουθώ τη συζήτηση και λέω ναι ως θεσμικό όργανο μπαίνουμε κάπως σε αχαρτογράφητα νερά. Και για να είμαι ειλικρινής, είμαι ευρωβουλευτής εδώ και μία εικοσαετία και μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει η συζήτηση για το εάν κάποιες χώρες μέλη τηρούν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρονολογείται από μακρού η συζήτηση αυτή και είναι ούτω ή άλλω άσχημο που καλούμαστε να συζητήσουμε τέτοια πράγματα. Και πράγματι στι χώρε μέλη υπήρξαν όντω φωνέ που ζήτησαν εάν κάποιος, μια κάποια χώρα δεν τηρεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να ρίχνουμε τόσα κονδύλια σε μια χώρα η οποία δεν τηρεί τις αξίες, τις οποίες βεβαίως κατά την ένταξή της έχει δεχτεί και συνυπογράψει. Ουδής υποχρεώνεται, εξαναγκάζεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερο, πρόκειται για μια κοινή σύμβαση την οποία έχουν υπογράψει όλες οι χώρες και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τηρήσουν τις σχετικές αρχές. Το ζήτημα τώρα του κράτους δικαίου, rule of law, καθορίζεται αρκετά σαφώ μέσα στι συνθήκε. Υπάρχουν και σχετικέ διαδικασίε που περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια. Εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακή Αναπτύξεω έχουμε προσπαθήσει ανέκαθεν να εξετάσουμε την μονομερή, επιβάρυνση της περιφερειακής πολιτικής και τη διασύνδεσή της με την αρχή τήρηση του κράτους δικαίου και έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει κάποιες βασικές αρχές δημοσιονομικού χαρακτήρα που να επιτρέπουν την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολισμού και τη διασύνδεσή του με το κράτος δικαίου. Ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει αυτό. Θα αποδειχθεί βεβαίως η ορθότητα του τρόπου αυτού συζήτηση με τις ε, διαβουλεύσεις που θα γίνουν. Ειδικά όμως για την δική μας Επιτροπή αξίζει τον κόπο να εγγύψουμε στο θέμα. Ότι υπάρχουν τώρα κανόνες για το αν κάποιος καταχράται τα χρήματα <clears throat> που πηγαίνουν στην ε, πολιτική περιφερειακή αναπτύξεως, αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε τώρα εδώ, διότι βεβαίως τότε μπορούν να πάψουν οι πληρωμές, να, ε, ζητηθούν, να ζητηθεί ανάκτηση των ε, οφειλωμένων κλπ. Χαίρομαι πολύ, άλλωστε που το ελεγκτικό συνέδριο βεβαιώνει ότι έχουν μειωθεί τα ποσοστά ασφάλματος στον τομέα της ε, περιφερειακής αναπτύξεως. Είναι πολύ θετικό σημάδι αυτό. Βεβαίως δεν πρόκειται ε, για το θέμα αυτό εδώ. Πρόκειται για το κράτος δικαίου. Και πράγματι ομολογώ ότι δεν έχω εξετάσει την γνωμοδότηση. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ προσεκτική και καθαρή δουλειά. Δεν ξέρω εάν η διαφθορά, η διαφθορά είναι ποινικό αδίκημα και βαρύ. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω λοιπόν αν η διαφθορά εμπίπτει σε θέματα κράτους δικαίου. Όταν λέει ο εισηγητής θα ήθελε να τα περιλάβει αυτά τα πράγματα στην ονομοδότησή ε, του, αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίες διαδικασίες όλων των χωρών μελών για να κάνουν τη σχετική έρευνα. Και αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο για την ώρα και θεωρώ ότι δεν υπάρχει και καμία απολύτως χώρα μέλος όπου να υπάρχει μηδενική διαφθορά. Δεν ξέρω λοιπόν αν πρέπει να συζητηθεί εδώ στην έκθεση αυτή, στην γνωμοδότηση αυτή, το θέμα της διαφθοράς ή αν πρέπει να συζητηθεί κάπου άλλο. Θεωρώ όμως ότι και ως Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξεως πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι χώρες μέλη οφείλουν να τηρούν το κράτος δικαίου εάν θέλουν να απολαμβάνουν την αλληλεγγύη των υπόλοιπων κρατών μελών. Θα παρακαλέσω λοιπόν κατά την σύνταξη της γνωμοδότησης που έχει και ε, μεγάλη πολιτική σημασία να προσεγγίσουμε το θέμα επικοδομητικά, να εξετάσουμε τι θέλουμε ακριβώς να αποτρέψουμε. δηλαδή να αποτρέψουμε τις χώρες από το να εγκαταλείψουν την οδό της αρετής, να σέβονται τις αρχές του κράτους δικαίου και να δούμε πώς μπορεί να προστατευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις, στα ενδεχόμενα αυτά. Οφείλουμε να διασαφίσουμε απολύτως τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για την πρώτη συζήτηση για το θέμα αυτό, λέει η Πρόεδρος. Είμαστε τώρα η αρμόδια επί ουσίας επιτροπή. Οι άλλες συναρμόδιες επιτροπές συντάσσουν τα νομοθετικά κείμενα. Αλλά για μας, για τη δική μας επιτροπή, το θέμα είναι σημαντικό, διότι πρόκειται για την διασύνδεση ανάμεσα στην στήριξη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή του κράτους δικαίου σε κάθε μια από τις χώρες μέλη. Αυτός ο σύνδεσμος θα πρέπει να είναι ισχυρό. Και νομίζω ότι εντάσσεται και στην προσπάθεια προστασία των συμφερόντων, όχι μόνο τη Ένωση, αλλά και των συμφερόντων του κάθε ενό πολίτου τη Ένωση. Γι' αυτό ζητούμε υπεύθυνη στάση πάντων σε ολόκληρο, το σύστημα. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Τόμασιτς, η οποία είναι σκιώδη συγγήτρια, έτσι δεν είναι. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά μόνο αν το ε, διοικητικό, νομικό και δικαστικό περιβάλλον στα κράτη-μέλη ε, υποστηρίζουν μια τέτοια ορθή χρήση. Ε, τα κράτη-μέλη ήδη έχουν την υποχρέωση να αποδεικνύουν ότι ισχύει ένας υγιής κανονιστικός μηχανισμός και ότι οι κανόνες εφαρμόζονται σωστά και ότι έχουν την απαραίτητη διοικητική ε, και θεσμική ικανότητα για μια επιτυχή χρηματοδότησή τους. Επιπλέον, οι όροι που τίθεται για τις πολιτικές αυτές ε, ευνοούν ε, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε τομείς όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν οικονομίες κλίμακος. Ε, ο κανόνα, το κράτος δικαίου είναι μια προϋπόθεση ε, για ένα κράτος ώστε να πάρει κοινωτική χρηματοδότηση και να αποδείξει ότι προστατεύονται ε, τα οικονομικά συμφέροντα της ε, Ένωσης. Αυτό αναφέρει η Κομισιόν σε μια ανακοίνωσή της του 2014. Συμφωνώ ότι η δικαιοσύνη ανεξάρτητα και αμερόληπτα ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά της και ότι θα πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες διαδικασίες και να εξασφαλίζεται το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι απαραίτητες σε μια ελάχιστη εγγύηση και εξασφαλίση κατά αυθαίρετων ε, αποφάσεων διαφόρων σωμάτων, οργάνων που μπορεί να ενεργούν, να έχουν σαν αποτέλεσμα να θυχτούν τα συμφέροντα της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμφωνώ όμως με την πρόταση του εισηγητή που θέλει να αφαιρέσει ε, από το Συμβούλιο τον ε, ρόλο στα πλαίσια αυτά. Δεν θα πρέπει να καταλήξουμε στο άλλο άκρο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, πολλές και διάφορες απόψεις, μεγάλη ποικιλία απόψεων. Θα ήθελα να καλέσω τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Budget να μας πει αν μπορεί να απαντήσει ας απαντήσει. Αν έχετε κάτι να εξηγήσετε, παρακαλώ να μας εξηγήσετε. Γιατί είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται και θα ήταν πολύ χρήσιμο να πάρουμε κάποιες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε εδώ λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνουν τα μέλη, ε, κύριοι Ευρωβουλευτέ, για την τόσο σημαντική αυτή η πρόταση τη Κομισιόν. Γιατί είναι σημαντική, Γιατί αποτελεί μέρο του πακέτου μας για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την επόμενη ε, περίοδο. Και είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι της νομοθεσίας, όπως πολύ σωστά είπε ο, ο Είναι μια ουσιαστική προϋπόθεση το κράτος δικαίου για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της Ένωσης στα κράτη-μέλη. Είναι πεπισμένη λοιπόν η Κομισιόν ότι ήταν απαραίτητο να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι υπάρχει ήδη αυτή η υποχρέωση ε, για τα κρατη να σέβονται το κράτος δικαίου, αλλά γενικευμένες ελλείψεις στον τομέα αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί η κανονική ε, ε, διοχέτευση κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα, ε, στα κράτη αυτά. Δεν πρόκειται για κυρώσει, δεν πρόκειται για τιμωρία, πρόκειται για την αποδοτικότητα. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε. Ο ορισμό. Ακούσαμε ε, αντικρουόμενες απόψεις από αυτού. Ε, δεν έχουμε όμως ξαναεφεύρει κάτι εδώ. Ο ορισμός προέρχεται από μια ανακοίνωση τη Κομισιόν και βασίζεται επίσης στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Και θα ήθελα να αναφερθώ στην ανακοίνωση ε, που έχει τίτλο «Το νέο πλαίσιο για το κράτος δικαίου». Ε, υπάρχουν επίσης αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του ε, Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής της Βενετίας κλπ. Ε, δεν προέρχεται από το πουθενά λοιπόν η έννοια αυτή. Υπάρχει ένας παγιωμένος ορισμός και επειδή πρόκειται για μια σημαντική πρόταση που θα έχει και δημοσιονομικές επιπτώσεις, ε, ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πολύ σωστό ορισμό του κράτους δικαίου. Περιλαμβάνει ο ορισμός αυτός την έννοια της νομιμότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, δημοκρατική και πλουριστική προσέγγιση για την υλοποίηση του νόμου, ε, ασφάλεια δικαίου, απαγόρευση της ε, αυθαιρεσίας, αποτελεσματική προστασία και ισότητα απέναντι στον νόμο. Έχουμε ένα περιεχόμενο λοιπόν. Το περιεχόμενο αυτό, όπως έλεγα, ε, γίνεται δεκτό ευρέως σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ. Για την διαφθορά, γιατί ε, τέθη αυτό το θέμα. Θεωρούμε ε, ότι το γεγονός ότι η διαφθορά δεν μπορεί να καταπολεμηθεί το θεωρούμε μάλλον το να μην μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η διαφθορά σε ένα κράτο μέλο είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό το λέμε στο άρθρο 3, όπου λέμε ότι τα μέτρα που θα πρέπει να πάρει ένα κράτο μέλο που υπάρχει κίνδυνο να επηρεάσουν τη σωστή προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση και αναφέρουμε στο γάμα μικρό, ε, αν δεν διερευνούν ή δεν διώκουν επαρκώς την απάτη ή τη διαφθορά. Υπάρχει λοιπόν σαφής αναφορά στη διαφθορά. Για τις εξουσίες και για τις αρμοδιότητες για τη χρήση των περιφερειακών ε, κονδυλίων. Υπάρχουν παρατυπίες, όλοι το ξέρουμε αυτό, ακόμα και απάτες. Και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν τελικά οικονομικές κυρώσεις σε επιμέρους, μονομένες περιπτώσεις, τις οποίες έχουμε ελέγξει και όπου έχει σαφώς ε, προσδιοριστεί ε, η παρατυπία, η απάτη και το ποσό για το οποίο πρόκειται. Εδώ Όμω, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Τι δίνει στην Κομισιόν αυτή η πρόταση. Δίνει στην ε, Κομισιόν την ε, εξουσία να αντιδράσει, όταν, όχι όταν υπάρχει μια μεμονωμένη παράβαση, αλλά όταν υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα, πέρα από ένα συγκεκριμένο έβριμα. Είναι ευρύτερο το πλαίσιο λοιπόν ε, και φυσικά πρέπει να σχετίζεται με το εύρος Τη γενικευμένη έλλειψη που διαπιστώνεται όσον αφορά το κράτος δικαίου. Ε, αυτό είναι, αυτή είναι η απάντηση ότι επιπλέον προσφέρει στην Κομισιόν η πρόταση αυτή. Επίσης, ε, αυτό σχετίζεται με την γενικότερη ε, αρμοδιότητα που έχει η Κομισιόν να προτείνει οριζόντιους κανόνες όπως τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς. Ε, η πρόταση αυτή λοιπόν καλύπτει όλα τα ταμεία και όλα τα κονδύλια και την έμεση και την άμεση διαχείριση και όχι μόνο την επιμερισμένη διαχείριση και γι' αυτό το προτείνουμε το σχέδιο αυτό σαν μια προϋπόθεση και μη ένα ε, συμπλήρωμα για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων για την αποτελεσματική προστασία. Γιατί έχουμε προτείνει μια συγκεκριμένη ε, διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Βασιζόμαστε σε ένα προηγούμενο που βασίζεται όχι στο κράτος δικαίου, αλλά στις οικονομικές προϋποθέσεις, στην καλή διακυβέρνηση, οι διαδικασίες που είναι συγκρίσιμες και που υπάρχουν και που εξασφαλίζουν ότι τα κράτη-μέλη ε, σέβονται τους οικονομικούς κανόνες υπάρχει η δυνατότητα και εκεί το Συμβούλιο να επέμβει με ειδική πλειοψηφία. Πιστεύουμε ότι έτσι υπάρχει σωστή ισορροπία. Αλλά προς το παρόν η Κομισιόν ακούει προσεκτικά όλες τις απόψεις σχετικά με το θέμα αυτό και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και έχει παρατηρήσει ότι μέχρι τώρα οι διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου έχουν υιοθετήσει διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν να τοποθετηθούμε και εμείς έως ότου δούμε ε, τι ε, θέσεις θα υιοθετήσετε τελικά αλλά για μένα δεν πρόκειται για καθαρή υλοποίηση του προϋπολογισμού εκ μέρου τη Κομισιόν. Δεν έχει νόημα αυτό, γιατί μιλάμε για περιπτώσεις γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου. Και μία απλή εφαρμοστική πράξη, στην περίπτωση αυτή, εκτελεστική πράξη εκ μέρους της Επιτροπής, θα ήταν πολύ light για μια τέτοια περίπτωση. Φυσικά περιμένουμε άμεση ενημέρωση από το Κοινοβούλιο μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Τέλος, για τους δικαιούχους αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί έχουμε ένα ειδικό άρθρο για τους δικαιούχους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποια από τα μέτρα αυτά μπορεί έμεσα να ζημιώσουν τους δικαιούχους. Έχουμε κάνει όμως ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να συμπεριλάβουμε σε αυτόν τον κανονισμό ό,τι είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση. Αν δείτε στο άρθρο 4.2, όχι μόνο προβλέπουμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι ανάλογα με το εύρος και το, τη σοβαρότητα των ελλείψεων, αλλά επίσης λέμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ποσοστό στο οποίο τα συμφέροντα της Ένωσης θίγονται από τις ελλείψεις αυτές και στη συνέχεια λέμε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γεγονός ότι υπόκειται στη διαδικασία αυτή ε, βάση του κράτους δικαίου, να χρησιμοποιήσουν αυτό αυτό σαν πρόσχημα για να μην καταβάλουν τα δέοντα στους τελικούς δικαιούχους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρεται μέσα σε ένα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σημαίνει ότι δίνει άμεσα το δικαίωμα σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πει δεν μπορεί να μου κόψει τη σύμβασή μου ή να την ε, ή να μην μου δώσει τα κονδύλια τα οποία δικαιούμαι, γιατί η κυβέρνηση ε, υπόκειται σε ένα τέτοιο μέτρο ε, που αφορά το κράτος δικαίου. Η κυβέρνηση δεν θα πάρει τη χρηματοδότηση, αλλά παρόλα αυτά θα έχει την υποχρέωση να ε, σεβαστεί τις συμβατικές υποχρεώσεις που ήδη έχει με τον τελικό δικαιούχο. Δεν είναι τέλεια η κατάσταση. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να επιλέξουμε μέτρα που δεν επηρεάζουν τον τελικό δικαιούχο και αν όχι προσπαθούμε να, θα, προσπαθήσουμε να εφαρμοστεί αυτό το άρθρο 4.2. Αυτή είναι μια πρώτη απόπειρα απάντησης. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βον Μίλτεμπιουρ θέλει να απαντήσει. Μάλιστα, πολύ σύντομα, γιατί πολλά έχουν ήδη υποθεί. Θα ήθελα μόνο την επιστρέψη τη προσοχή στο γεγονό ότι πρόκειται για μια νομοθετική γνωμοδότηση. Επομένω, είναι λογικό να υπάρξει και μια διάσταση απόψεων. Όμω, είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η γνωμοδότηση και να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συμβαστικό κείμενο, γιατί πουθενά αλλού δεν θα ακουστεί η γνώμη μα. Αν απλώ το απορρίψουμε και δεν υπάρξει ένα κείμενο συμβασμό, θα έχουμε δύο καθήλυνα αρμόδιε επιτροπέ που δεν θα λάβουν υπόψη τα δικά μα σχόλια. Και μια μικρή μνήμα στα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα ενισχύσουμε την πρόταση αυτή εάν αφαιρέσουμε όλα τα στοιχεία που κατά το μάλλον ή τον ε, συνδέονται με τη διαδικασία του άρθρου 7. Γιατί πραγματικό μέλημα εδώ είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση. Δεν είναι πρόταση που άπεται του κράτου δικαίου. Ε, μία αποδυναμωμένη δηλαδή εκδοχή της διαδικασίας του άρθρου 7. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, και έχουμε και την νομοδότηση της κυρίας Β, από το ε, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στην Φλωρεντία, ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, ότι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά στηρίζει την πρόταση αυτή στα άρθρα που έχουν να κάνουν με την δημοσιονομική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να επιμείνουν σε αυτά τα άρθρα και μόνο, το 322 και 317 που αφορούν την εκτέλεση του προπολογισμού. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης αναφέρεται και στην μελέτη, έχει ξεκάθαρη αρμοδιότητα. Δεν χρειάζεται λοιπόν εκεί να παρεμβαίνει το Συμβούλιο, γιατί αυτό μάλλον θα περιπλέξει τα πράγματα. Φυσικά, πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ενημερώσει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, αλλά είναι δική της αρμοδιότητα και ευθύνη. Αυτά είχα να πω και προσβλέπω στη συνέχιση των συνομιλιών. Σας ευχαριστούμε πολύ καθώς οι καθήλυν αρμόδιες επιτροπές budget και κοντ θα ψηφίσουν για αυτή την νομοθετική έκθεση στο τε, στα τέλη Νοεμβρίου, εμείς θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 15 Νοεμβρίου το αργότερο. Γι' αυτό και προτείνω μια προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 19 Οκτωβρίου το μεσημέρι, ημέρα Παρασκευή. 19 Οκτωβρίου λοιπόν. Και σίγουρα και η συζήτηση μεταξύ των σχεδόν εισηγητών θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ας συνεχίσουμε. Να σας επενθυμίσω ότι έχετε λάβει μέσω mail τις αποφάσεις των συντονιστών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης. Μπορούμε να εγκρίνουμε τις αποφάσεις. Υπάρχουν σχόλια. Α, ναι. Ε, και η απόφαση για την συνάντηση της 27ης έχει κυκλοφορήσει. Ωραία, συμφωνούμε και εγκρίνουμε. Υπό τα διάφορα υπάρχει κάτι. Όχι. Η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα στις 15 Οκτωβρίου το απόγευμα από τις 3 έως τις 6.30. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Η Προέδρος ευχαριστεί ευγενικά τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ για την ε, συμμετοχή σας και την υπομονή σας σήμερα το απόγευμα. Γεια σας.